Να ξεκινήσουμε αγαπητοί συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω στη συνεδρίαση αυτή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Ε, σημείο 1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Σε ό,τι αφορά τα σημεία το και 7 έχει προταθεί να συζητηθούν μετά το 3. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις και θεωρώ ότι εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε η ημερήσια διάταξη. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ανακοινώσεις του πρωί, το σημείο 2, δεν έχω να σας πω κάτι. Επομένως, μπορούμε να προχωρήσουμε ευθύς αμέσως στο σημείο 3. που είναι η παρουσίαση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του θέματος ε, της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου και των κανόνων της Ένωσης στον τομέα της ε, αστικής ε, δικαιοσύνης και του Εθνούς Ιδιωτικού Δικαίου. Από τις 30 Μαρτίου του 2019 και από τις 12 η χώρα του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι τρίτη χώρα βέβαια με την επιφύλαξη άλλων δυνητικών πολιτικών εξελίξεων. Επειδή υπάρχουν αβεβαιότητες και ασάφεις ό,τι αφορά την κύρωση της συμφωνής αποχώρησης, θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν ακριβώς ποιες είναι οι νομικές επιπτώσεις που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Είναι σημαντικό να προετοιμαστούν ε, για την αποχώρηση του Βασιλείου οι εθνικές αρχές, οι ενωσιακές αρχές αλλά και οι ιδιωτικοί φορείς. Με την επιφύλαξη λοιπόν της σύναψης ε, της συμφωνίας αυτής και της επικύρωσής της και της μεταβατικής περίοδου θα πάψουν να ισχύουν οι κανόνες της Ένωσης για το Ηνωμένο Βασίλειο ό,τι αφορά ε, το αστικό δίκαιο και το διεθνές ιδιωτικό δίκαιο και αυτό αφορά ιδίω τη διεθνή δικαιοδοσία, αναγνώριση, επιβολή και ειδικών διαδικασιών, δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Καλέσαμε λοιπόν για όλους αυτούς τους λόγους την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας ε, παρουσιάσει τις επιπτώσεις της αποχώρησης. Νομίζω ότι έχουμε εδώ τον κύριο Αντρέα Στάιν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 οι άμεσες επιπτώσεις ε, μιας ε, εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία. Δεν μιλάω για τις ε, συνέπειες της επικύρωσης συμφωνίας αποχώρησης, γιατί με αυτές ουσιαστικά για τη, για τη μεταβατική περίοδο παραμένουν σε ισχύ κανένας ένωση. Μιλάω για τις άμεσες επιπτώσεις ενός no deal. Άμεσες δε επιπτώσεις όταν λέω αποκλείω και εξαιρώ και το θέμα των μελλοντικών σχέσεων της Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία. Άρα, ουσιαστικά θα σας πω τι πρόκειται να συμβεί σε περίπτωση που αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη Μαρτίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης. όπως είπατε και εσείς σε αυτή την περίπτωση και επειδή στον τομέα της ε, αστικής ε, δικαστικής συνεργασίας ε, ε, βασιζόμαστε στους κανονισμούς ε, που είναι νομικά μέσα άμεσα εφαρμοστέα. Οι συνέπειες ενός Brexit χωρίς συμφωνία είναι πως όλα αυτά τα νομικά μέσα από τη μία μέρα στην άλλη πάβουν να εφαρμόζονται, πάβουν να ισχύουν σε ό,τι αφορά το νομένο Βασίλειο. θα σας αναφέρω δύο-τρία θέματα, αλλά το βασικό θέμα είναι ότι δεν θα εφαρμόσετε πλέον για το Ηνωμένο Βασίλειο ε, η ενωσιακή δομοθεσία από την ημερομηνία αποχώρησή του και μετά, που σημαίνει ότι θα υπάρξει ένα νομικό κενό λόγω της μη ε, εφαρμοσμότητας του ενωσιακού δικαίου. Και αυτό το κενό πρέπει να καλυφθείται από εθνικό δίκαιο που θα εφαρμόζεται αντί του ε, ενωσιακού και αν υπάρχουν διεθνείς, διεθνείς συμφωνίες, στις οποίες είναι συμβαλόμενα μέρη η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο θα ισχύουν. Θα σας πει η Πατρίσα Ντελούκα, η Συνόδο που είναι εδώ, κάποια πράγματα για αυτές τις διεθνεί συμφωνίε. Για κάποια θέματα τώρα πιο συγκεκριμένα, να ξεκινήσω με το λιγότερο προβληματικό, που είναι η σύγκρουση των ε, εφαρμοστέων κανόνων δικαίου. Όταν ε, ε, μιλάω γι' αυτό, εννοώ τους κανονισμούς Ρώμη 1 και 2 που βεβαίω και θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται ενώ με των δικαστηρίων των 27 δεν υπάρχει αμοιβαιότητα σε ό,τι αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο. Γνωρίζουμε επίσης από τις ε, ανακοινώσεις του Ρωμένου Βασιλείου ότι σκοπεύει, προτίθεται να συνεχίσει να εφαρμόζει τις ε, δύο αυτές, ε, τα δύο, τους δύο κανονισμούς Άρα σε ό,τι αφορά τους εφαρμοστέους κανόνες, εκεί δεν θα έχουμε μάλλον πρόβλημα, γιατί και από τις δυο πλευρές θα συνεχίσουν τα δικαστήρια να εφαρμόζουν ε, τους ίδιους κανόνες. Τώρα, σε ό,τι αφορά του κανόνε διεθνού δικαιοδοσία που εναρμονίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά αστικά εμπορικά ζητήματα, ζητήματα οικογενειακού δικαίου και ζητήματα πτώχευση ε, και αφαιρεγκαιότητα. Εδώ πρέπει να κάνουμε μία διάκριση. Έχουμε δύο διαφορετικές καταστάσεις. Η απλή η περίπτωση είναι όλες οι δικαστικές διαδικασίες οι οποίες ε, κινούν από την μερμηνέα αναχώρηση και μετά νέες δηλαδή διαφορές ε, και δικαστικές διαδικασίες μετά τον Brexit δεν θα εφαρμόζεται σαφώς εδώ το κοινωτικό κεκτημένο που σημαίνει ότι τα δικαστήρια των 27 χωρών δεν θα εφαρμόζουν αυτά τα νομικά μέσα παρά μόνον εφόσον ρητό αναφέρει αυτό το νομικό μέσο ότι εφαρμόζεται ενωσιακό σε ό,τι αφορά τους εναγωμένους στο Ενωμένο Βασίλειο και το έχουμε αυτό στο κανονισμό Βρυξέλλες 1 σε κατανοητικά ζητήματα που λέει ότι οι κανόνες αυτοί εξακολουθούν να ισχύουν ανεξαρτήτως ε, της ε, έδρας ε, του καθού, του εναγωμένου. Μπορεί να είναι στο Βασίλειο, μπορεί να είναι στην Ευρωπαϊκή Θα συνεχίσει να ισχύει ο κανονισμός Βρυξέλλης 1. Αλλά ε, πέραν των συγκεκριμένων αυτών περιπτώσεων, τα 27 ε, κράτη-μέλη και τα δικαστές δεν θα εφαρμόζουν τις Βρυξέλλης 1, παραδείγματο χάρη, αλλά ε, τους εθνικούς κανόνες για διεθνή δικαιοδοσία, εκτό αν υπάρχει διεθνή συμφωνία ή σύμβαση που να καλύπτει αυτά τα ζητήματα. Δεύτερο σενάριο διαφορές, διδεσυνομικές διαμάχε, οι οποίε εκκρεμούν. Έχουν ξεκινήσει δηλαδή πριν το Brexit, αλλά εξακολουθούν ε, να μην έχουν ολοκληρωθεί ε, και μετά το Brexit. Από τη σκοπιά των 27, οι κανόνες θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται για την προστασία των νομικών, θεμητών νομικών προσδοκιών ε, των μερών, των διαδίκων που ξεκίνησαν τη διαδικασία και από το guidance note, αυτή το σημείωμα, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο προτίθεται να κάνει το ίδιο αυτό, απορρέει. Δηλαδή για τους σκοπούς διεθνούς δικαιοδοσίας ε, οι διαδικασίες αυτές δικασίες θα συνεχίζουν να, να ε, τηρούν και να σέβονται τους κανόνες που σέβονταν όταν ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Ό,τι αφορά τα αναγνώριση και την επιβολή, εδώ τα πράγματα περιπλέκονται κατά τη και γίνονται λίγο πιο προβληματικά για τους διαδίκους, διότι εδώ μιλάμε για θέματα αμοιβαιότητας. Συνήθως σε διμερείς συμφωνίες μεταξύ χωρών υπάρχει προνομιακή αναγνώριση αν έχει την ίδια αντιμετώπιση και μεταχείριση και από την άλλη χώρα. Η αρχή εδώ είναι απλή επίσης για τις διαδικασίες οι οποίες ξεκινούν και εδώ μιλώ για διαδικασίες επιβολής που ξεκινούν από την ημερομηνία του Brexit και μετά ή συνεχίζονται από τη μέρα του Brexit και μετά. Δηλαδή, μπορεί η ετοιμιγορία να έχει ε, δημοσιοποιηθεί πριν, αλλά η επιβολή της γίνεται μετά. Και οι προνομικοί κανόνες για την αναγνώριση και την επιβολή δεν εφαρμόζονται πλέον που σημαίνει ότι ακόμη και αν μια απόφαση έχει ε, δοθεί πριν την ημερομηνία του Brexit και ακόμη και επιστραφή στις αρχές επιβολής νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου για πριν την ημερομηνία του Brexit ε, για να επιβληθεί, να εφαρμοστεί η απόφαση, δεν έχει εφαρμοστεί τη στιγμή της αποχώρησης, άρα δεν συνεχίζουν οι κανόνες να εφαρμόζονται για αυτές τις διαδικασίες επιβολής πολύ ξεκάθαρη τομή. Μία μόνη εξαίρεση στον κανόνα αυτό. Δηλαδή όταν μια απόφαση έχει ήδη πάρει εκτελεστική, ε, εκτελεστικό χαρακτήρα, είναι εξακβάτορο όπως λέμε. Αν έχει δηλαδή υπάρξει δήλωση εφαρμοσιμότητας για τη Γαλλία, παραδείγματος χάρη με την ημερομηνία του Brexit, σε αυτή την περίπτωση και για πολλές περιπτώσεις του κεκτημένου δεν υπάρχει απέτηση εξ εκβάτορ. Αλλά για παλαιότερες ε, εμπορικές υποθέσεις ε, και υπό το Βρυξέλλες 2 που δεν είχε καταργήσει εντελώς το εξεκβάτορ. Υπάρχουν περιπτώσεις που για αστικές ή εμπορικές υποθέσεις παραλαμβάνω χρειάζεται δήλωση εφαρμοσιμότητας ε, ή επιβολής στη χώρα που θέλουμε να γίνει επιβολή. Αν έχουμε λοιπόν μία απόφαση για το Ηνωμένο Βασίλειο και έχει πει το Γαλλικό Δικαστήριο ότι αυτή η απόφαση ε, εκτελείται ε, στο γαλλικό έδαφος πριν την μερνία του Brexit, δεν καταλαβαίνουμε γιατί η εθνική αυτή γαλλική απόφαση που βασίζεται στο κεκτημένο, κατανοητό αυτό, γιατί να μην πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται στο γαλλικό έδαφος και μετά το Brexit. Αλλά αυτή είναι η μόνη μικρή σχετικά εξαίρεση που μπορέσαμε να σκεφτούμε. Εκεί όπου δηλαδή οι κανόνε αναγνώριση και επιβόληση εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ημερομηνία του Brexit. όλε τι άλλε περιπτώσει, ακόμη και αν η απόφαση έχει ε, πάρθει πριν και η ημερομηνία επιβολή είναι μετά, πάβουν να ισχύουν οι κανόνε από τη μέρα τη αποχώρηση και μετά. Άρα οι αποφάσεις θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να εφαρμόζονται, να επιβάλλονται ε, στη βάση του εθνικού δικαίου. οι δικαστικές διαδικασίες έχουν εθνικούς κανόνες ε, για την αναγνώριση και την επιβολή ξένων αποφάσεων και αυτό θα ισχύει για τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αποφάσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τον Brexit. Τρίτο θέμα. Ειδικέ ενωσιακέ διαδικασίες. Όπως ξέρετε, δημιουργήσαμε κάποιες ειδικές διαδικασίες, παραδείγματος χάρη για μικρές αξιώσεις, το small claims ή το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Πληρωμών. Η σχετική διαδικασία θεσπίζει συγκεκριμένα πράγματα που είναι αναρμονισμένα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμπληρώνονται με ειδικού κανόνες περί αναγνώρισης και επιβολής ε, εφαρμογής αυτών των αποφάσεων που απορρέουν από τέτοιε διαδικασίε. Πολύ σύντομα ε, μπορώ να τα πω για αυτό το θέμα, γιατί οι αρχέ που άπτονται τη δικαιοδοσία και τη αναγνώριση και επιβολή τι νομοθεσίε συγκεκριμένε αυτέ, ειδικέ ενωσικέ διαδικασίε, είναι οι ίδιε ακριβώ με αυτέ που περιέγραψα προηγουμένω για τι τακτικέ ε, μη ειδικέ ενωσικέ διαδικασίε. Άρα θα εφαρμοστούν εδώ οι ίδιε αρχέ. Να πω δύο λόγια και για του ειδικούς μηχανισμούς δικαστικής συνεργασίας στο πλαίσιο του και εκτιμένου, του νοσιακού εκτιμένου. Οι αρχέ των κρατών μελών, τα δικαστήρια, κεντρικές αρχές κτλ. κτλ παρέχουν δικαστική συνδρομή και συνεργασία σε ό,τι αφορά την επίδοση εγγράφων ε, ε της καταθέσεις, της ε, ε συνεργασίας με ξένες αρχές στην περίπτωση αρπαγής παιδιών και τα του κανονισμού Βρυξέλλες 2. Εδώ τι γίνεται. Έχουμε ένα πολύ ξεκάθαρο κανόνα που λέει ότι αυτοί οι μηχανισμοί συνεργασίας πάβουν να, ισχύουν την μέρα αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Δηλαδή ακόμη και αιτήματα τα οποία είχαν γίνει πριν την ημερομηνία αποχώρηση για την επίδοση ενό εγγράφου σε ό,τι αφορά τη συνεργασία για την πέτωση αρπαγή ενό παιδιού, δεν θα συνεχίσουν ε, να εμπίπτουν ε, στην ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μετά δε την αποχώρηση δεν θα μπορεί καν να ξεκινήσει μια νέα υπόθεση δυνάμεων με, με βάση τους νοσιακούς κανόνες. Άρα θα πρέπει είτε εθνικό δίκαιο είτε διεθνή συμβάση να καλύψουν αυτό το νομικό κενό. Έχουμε την Σύμβαση της Χάγης για την Αρπαγή των Παιδιών, που προβλέπει συνεργασία μεταξύ των κεντρικών αρχών. Και επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο είναι συμβαλλόμενο μέρο στη σύμβαση, όπω και όλα τα άλλα κράτη-μέλη τη Ένωση, η συνεργασία μπορεί να συνεχιστεί. Άρα εδώ οι συμβάσει διεθνεί έχουν το ρόλο του. Σε ό,τι αφορά όμω το ενωσιακό κεκτημένο, πάβει να ισχύει. Τέλο, πολύ σύντομα, δημόσια έγγραφα. Έχουμε τον κανονισμό για τα δημόσια έγγραφα που απλουστεύει τις διατυπώσεις ε, για την ε, παρουσίαση των ε, δημοσίων εγγράφων σε ένα τρίτο κράτος με την κατάργηση της υποχρέωσης για την επισημείωση της Χάγης. Και αυτό ισχύει για οποιαδήποτε έγγραφο θα κατά του πότε εκπονήθηκε. Πριν την αποχώρηση, η απλούστευση αυτή, η δυνάμη του κανονισμού για τα δημόσια έγγραφα πάδινα ισχύει. Και το τελευταίο που ήθελα να πω είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστικό ε, Δίκτυο και το e-justice, η πύλη αυτή. Ξαφής διαχωριστική γράμμη. Από την ημέρα αποχώρησης χωρίς συμφωνία το ε, Ηνωμένο Βασίλειο πάβει είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου και δεν θα υπάρχουν πληροφορίες ε, στο e-justice ε, ε, από τη στιγμή εκείνη και μετά. Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς συμβάσεις, είπα ότι είναι μια λύση γι' αυτό. το κενό που και θα δώσω το λόγο στην κυρία Λούκα, τη συνάδελφό μου. Ευχαριστούμε, ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Κοιτάξτε, ε, δεν γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι σε ορισμένες ε, περιπτώσεις, σε διεθνείς συμβάσεις, όπως ε, αυτές ε, που έχουν που υπάρχουν στο διεθνές δίκαιο, ότι τέτοιου είδου συμβάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μια περίπτωση για να μπορούμε να έχουμε κάποια λύση. Βέβαια, Στη σύμβαση δεν αναφέρονται όλα τα θέματα τα οποία εξετάζονται σήμερα στα πλαίσια του ενωσιακού δικαίου. Όσον αφορά το ενωσιακό εργαλείο, ε, το οποίο ισχύει, παραδείγματο κάνει κανονισμό Βρυξέλλε 1, υπάρχει μια σύμβαση η οποία ε, μπορούν να υπάρχει μια βάση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έκτακτη, λύση έκτακτης ανάγκης ε, είναι η απόφαση αυτή που έχει λάβει και το δικαστήριο. Πάντως αυτή είναι μόνο μια ενωσιακή σύμβαση που σημαίνει ότι έχει υπογραφεί και κυρωθεί μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η κύρωση δεσμεύει όλα τα κράτη-μέλη. Βέβαια, καθώς ε, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ε, συμμετάσχει στην ε, διπλωματική συνεδρίαση που έχει εγκρίνει αυτή την σύμβαση, έχει τη δυνατότητα και αυτό να επικυρώσει. Και αυτό έχει ήδη γίνει τέλη Δεκεμβρίου, τέθη σε ισχύ τον Απρίλη, έτσι ώστε να αποφευθούν ή δυνατόν οποιαδήποτε κενά ε, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία παρεμφερή κατάσταση βρίσκουμε και στην ε, υποχρέωση διατήρησης. Εδώ έχουμε ε, την ε, Σύμβαση για την ε, Διατροφή για τα Παιδιά και για τις Συζύγους. Εδώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη εκ των προτέρων κυρώσει αυτή τη σύμβαση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Απριλίου. Υπάρχουν και άλλες συμβάσεις όπου το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τις δικές του συμβάσεις, την 95 και την 96, 96 συγκεκριμένα, αφορά την προστασία των παιδιών. Η προηγούμενη αφορούσε θέματα απαγωγή του. Αυτέ οι δύο συμβάσει ε, είναι οι ε, προκάτοχοι ε, του κανονισμού Βρυξέλλες 2α. Βέβαια υπάρχουν άλλοι τομείς όπου η κατάσταση είναι πολύ πιο περίπλοκη, παραδείγματο χάρη όσον αφορά την αναγνώριση ε, των διαζυγίων. Αυτό καλύπτεται από την Σύμβαση 2α και επίσης και από τη Σύμβαση 90-70 ε, που ε, άπτεται της αναγνώρισης των διαζυγίων. Εδώ όμως Υπάρχει αυτό το 12 το οποίο επίσης ε, καλύπτει και το ε, Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει λοιπόν ε, περιορισμένη δυνατότητα για να ισχύει κάποια λύση έκτακτης ανάγκης και τα κράτη-μέλη ε, που θέλουν να είναι μέλη αυτής της σύμβασης. Αυτό θα πρέπει ε, να ε, προταθεί και να καλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την δικαστική συνεργασία, η σύμβαση 2α επί του ιδίου θέματος μπορεί και αυτή να χρησιμοποιηθεί και εδώ όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει ε, να ε, προσχωρήσουν στην Σύμβαση για την Παροχή Υπηρεσιών. Βέβαια, αυτή η σύμβαση δεν έχει ακόμα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη έχουν τοποθετηθεί εκτός από την Αυστρία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία Αυτές λοιπόν είναι οι λύσεις και οι δυνατότητες που υπάρχουν και θα ήθελα να προσθέσω ότι υπάρχουν και διμερείς συμφωνίες, ε, κυρίως ε, από τις ε, δεκαετίες του 20 και του 30 που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως και αυτά βέβαια ήταν πριν συσταθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι βέβαια αυτές οι συμβάσεις είναι ξεπερασμένες από το ενωσιακό δίκαιο και ως εκ τούτου ε, δεν μπορούν να ισχύουν πλέον για να ρυθμίζουν τις σχέσεις ανάμεσα στον Ηνωμένο Βασίλειο και τα κράτη-μέλη. Ε, και προφανώς ε, θα πρέπει να υπάρχουν και νέες συμφωνίες οι οποίες ήδη καλύπτονται από το ενωσιακό δίκαιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Much. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν ε, κάποιος από τα μέλη θέλει να κάνει μία ερώτηση στην ε, Επιτροπή. Από ό,τι βλέπω, ε, κανείς δεν θέλει κάποια ερώτηση. Ταντέους, σύντομα σας παρακαλώ αν έχει την καλοσύνη. Ε, πράγματι θα είμαι σύντομος, ε, μια πάρα πολύ σύντομη ερώτηση και πολύ ε, συγκεκριμένη ερώτηση που αφορά στην συνεργασία μετά το Brexit. Πρώτα απ' όλα, σε σχέση με την εφαρμογή της συνθήκης της Χάγης. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό τόσο το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα κρατημέλη έχουν προσχωρήσει σε αυτήν την σύμβαση, όμως έχουμε ένα πρόβλημα στο να ολοκληρωθεί ε, η διαχειριστική, διοικητική μάλλον συμφωνία η οποία ισχύει τώρα και αυτό ε, προσπαθώντας ε, να επιτύχουμε να αποκτήσουμε τις διευθύνσεις ατόμων που οφείλουν διατροφές. Ίσως τελικά μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτό το έγγραφο. Και κάτι άλλο. Έχει σχέση με το ότι η συνεργασία δεν θα καλύπτει λιγότερο επίσημους ε, ε, φορείς Νομίζω αυτό πλέον δεν θα ισχύει για τους Βρετανούς δικαστές και αυτό ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη μετρατική περίοδο, όπου θα είναι όμως απαραίτητο να υπάρχει συνεργασία, γιατί ε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε σχεδόν από το μηδέν. Ίσως ε, λοιπόν ε, να πρέπει να σκεφτούμε να αφήσουμε για κάποιο χρονικό διάστημα τους εκπροσώπους του Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτά τα δίκτυα. Εντάξει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει κάποιο σχόλιο να κάνει. Παρακαλώ σύντομα, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος για το πρώτο σημείο που αναφέρθηκε και για τους περίπλοκους μηχανισμούς και για το καθεστώς διατήρησης της εθνικότητας, θα υπάρχει ένα τμήμα που πρέπει να πληρώσουμε όλοι και το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί, που δεν θα είναι πλέον τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να υπάρχουν ανεπιθύμητες παρενέργειες, διότι η συνεργασία με τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ πιο ε, καλά οργανωμένη σε σχέση με τη Σύμβαση της Χάγης. Δεν θέλουμε όλα αυτά να γίνουν παγιωμένη κατάσταση και στο απότερο μέλλον. Δεν έχουμε ακόμα απαντήσει το θέμα της μελλοντική μας σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο, ούτε το καλύψαμε στην παρουσίασή μα σήμερα. Πάντως, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο υπάρχει ε, πρόβλημα και με τη σύμβαση που, του δικαστικού δικτύου που δεν θα ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει δυνατότητα σε κάποιες περιπτώσεις να προσκαλούνται τρίτες χώρες στο δικαστικό δίκτυο για να ε, λυθούν θέματα αν χρειαστεί, είναι ένα έκτακτο μέτρο. Και δεν ξέρουμε αν είναι η καταλληλότερη σχέση που θέλουμε να δημορφώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τον Brexit. Πάντω η αρχή ότι δεν μπορούν πλέον να είναι μέλο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού ε, Δικτύου είναι μια αναπόφευκτη συνέπεια του Brexit χωρί συμφωνία. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθε σήμερα και σα ευχαριστώ και για αυτή την παρουσίαση. Και θα συνεχίσουμε με το 8. Την σύναψη διαθεσμικών διαπραγματεύσεων και τα μη δεσμευτικά κριτήρια για την εφαρμογή των άρθρων 290 και 291 της συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. TFU. Οι συνδιαπραγματευτές είναι ο κύριος Σάγερ και ο κύριος Κόρμπετ. Δυστυχώς δεν ήρθαν. Ζητούν συγγνώμη. Μου ζήτησαν ωστόσο να σας διαβάσω το μήνυμά τους το μήνυμα του κυρίου Σάγερ συγκεκριμένα. Και ξεκινάω. στι 9 Ιουνίου 2016 η διάσκεψη των Προέδρων ανέθεσε σε μένα και τον κύριο Ρίτσαρτ Κόρμπετ εντολή για να διαπραγματευτούμε εκ μέρου του Κοινοβουλίου μη δεσμευτικά κριτήρια για τι κατεξουσιοδότηση και εφαρμοστικέ πράξει βάσει των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του εδαφείου 28 Τη Διαθεσμική Συμφωνία για την Καλύτερη Νομοθεσία του 2016. Η εντολή ήταν να διαπραγματευτούμε βάσει των κριτηρίων που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου του 2014 για τις καθεξουσιοδότηση και εφαρμοστικές πράξεις. Ήμουν ε, υπεύθυνο για το ντοσχέ αυτό. Ε, οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο επισήμως ξεκίνησαν επί της εστονική Προεδρίας στι 12 Σεπτεμβρίου 2017. Επιπλέον συναντριάσεις οργανώθηκαν επί Βουλγαρικής και Αυστριακής Προεδρίας και καταλήξαμε σε καταρχήν συμφωνία για τα κοινά κριτήρια στις 29 Νοεμβρίου 2018. Είμαι ικανοποιημένο που η συμφωνία που επιτύχαμε ε, είναι αυτή τη μορφή, γιατί θεωρώ ότι τα μη δεσμευτικά κριτήρια θα βοηθήσουν να υπερπηδήσουμε εμπόδια, τα οποία έχουν ε, αναδυθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα για τις ε, νομοθετικές μας διαπραγματεύσεις που μπορεί αλλιώς να μπλοκαριστούν στο επίπεδο των κατεξοδότηση και εφαρμοστικών πράξεων. Τώρα, τα κριτήρια αυτά της ε, οριοθέτησης θα βοηθήσουν τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών και θα επιτρέψουν να είναι καλύτερη και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πολίτες. Τα μη δεσμευτικά κριτήρια είναι μια μορφή μιας ε, ανεξάρτητης συμφωνίας και θα δημοσιευτούν στην ε, σειρά γάμα της επίσημης εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να έχουν πρόσβαση όλοι. Ε, σε ό,τι αφορά τη χρήση των κατεξουσιοδότητων εξουσιοδότηση και εφαρμοστικών πράξεων στον τομέα του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορετικέ θέσει των τριών θεσμικών οργάνων επί του θέματο, συμφωνήθηκε να μην γίνει συγκεκριμένη μνήμα στο ζήτημα αυτό, αλλά να ισχύσουν οι γενικέ αρχέ των κριτηρίων. Το κείμενο των μη δεσμευτικών κριτηρίων έχει τώρα υποβληθεί στη διάσκεψη των Προέδρων για να το εγκρίνουν και από πολιτικής σκοπιάς. Οπότε, αυτά μπορώ να σας πω εκ μέρους του κυρίου Σάγκερ. Δεν έχω μήνυμα από τον κύριο Κόρμπετ όμως. Έχει κανείς κάποιο σχόλιο από το θέμα τους. Δεν μοιάζει να υπάρχει κανείς που να έχει σχόλιο από το θέμα τους. Θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Uh, uh, Πριν ψηφίσουμε στις 15 και 40 θα συνεχίσουμε με το σημείο 7 την ενημέρωση της Επιτροπής μας για τις διαπραγματεύσεις βάσει του άρθρου 69 ε, εδάφιο 3. για την προσαρμογή κάποιων νομικών πράξεων που ασχολούνται με την εφαρμογή της ρυθμιστικής διαδικασίας και τη λογοδοσία βάσει των άρθρων 290 και 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, TFU. αυτή ε, στιγμή εισηγητή πάλι είναι ο κύριο Σάγερ και δεν βρίσκεται εδώ όπω προείπα. Ε, θα σας διαβάσω το μήνυμά του. Τα τρία θεσμικά όργανα στις 12 Φεβρουαρίου 2019 πέτυχαν μια προσωρινή συμφωνία για να ευθυγραμμίσουν τις πράξεις ε, προ τη συνθήκη τη Λισαβόνα, που είναι 64 στον αριθμό, για τη χρήση τη ρυθμιστική διαδικασία με λογοδοσία βάσει των άρθρων 290 και 291 τη συνθήκη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την εφαρμογή της Διαθεσμικής Συμφωνίας του 2016 για την καλύτερη νομοθεσία στον τομέα της έγκαιρης ευθυγράμμισης βάση της οποίας τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δίνουν υψηλή προτεραιότητα σε όλες τις βασικές πράξεις και θα πρέπει όλες αυτές να υπόκεινται στην ρυθμιστική διαδικασία με λογοδοσία. Η δουλειά μας δεν ήταν απλή, καθώς τα τρία θεσμικά όργανα βλέπουν κάποιους στόχους από τελείως διαφορετική σκοπιά. Όμως έχουμε δείξει στους πολίτες ότι μπορούμε να υπερπηδήσουμε τέτοια διαθεσμικά, τέτοια μάλλον θεσμικά συμφέροντα προς όφελος μιας εύρυθμης και ε, εύρωστης Ευρώπης. Δεν έχει τελειώσει όμως η δουλειά μας. Η ευθυγράμμιση των ε, εναπομεινάσεων των εναπομεινασών 104, 104 πράξεων ε, παραμένει ε, κάτι που θα μας απασχολήσει και θα χρειαστούν διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ όλους τους χιόδους εισηγητές για τη συμμετοχή τους στις συναντήσεις μας. Εξ αρχής ήταν πολύ συνεργάσιμοι και αυτό επέτρεψε να ε, δείξουμε ότι το Κοινοβούλιο έχει μια ισχυρή θέση στις διαθεσμικές διαπραγματεύσεις. Σας παρακαλώ να υποστηρίξετε την προσωρινή συμφωνία ε, ψηφίζοντας υπέρ. Θα κάνουμε τώρα μια μικρή διακοπή ω τι 15.40 για να αρχίσουμε ακριβώς την ώρα που έχουμε γράψει και στην ημερήσια διάταξη και έχουμε αναγγείλει. Uh, Συνάδελφοι, να συνεχίσουμε με τις ψηφοφορίες. Ελπίζω ότι όλοι έχετε εισαγάγει την κάρτα σας στην ε, κατάλληλη θέση. Περνάμε στο σημείο 7. Νομοθετική διαδικασία ρυθμιστική διαδικασία με πράξεις λογοδοσίας. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Shall we wait for him? Mr. Anderson is not looking. No. No. yes, we have it. So, okay, let's close it it has Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια στον κύριο Σάιερ. the legal on... Σημείο 1 για την η έδρα για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Ολοκληρώνεται. 19.00. Uh, Συγχαρητήρια στον εισηγητή, τον κύριο Λεμπρετών. Και άλλη έκθεση Λεμπρετών, νομική βάση για την πρόθεση των καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οδικών οχημάτων. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και πάλι συγχαρητήρια στον εισηγητή. Μετά αναφορά του Πιέρ Παόλο Βόλπε, άρχεται η ψηφοφορία. Close 19 ε, εγκρίνεται 19.00. Κυρία Ρέγνερ. Um, um, Ευχαριστώ. Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία της έκθεσης ΖΙΦΚΑ, εκ μέρου ε, του σκιώδη συγγετή συγκεκριμένα, τη κυρίας Γκούτελαντ και εξ ονόματό μου, θέλω να πω ότι αυτή η οδηγία εντάσσεται στο πακέτο για το εταιρικό δίκαιο. Περιλαμβάνει και μια συνεκτική πρόταση για μια νέα οδηγία για διασυνοριακές συγχωνεύσεις, διαιρέσεις ε, και χαιρόμαστε που στην οδηγία για τα ψηφιακά εργαλεία περιλαμβάνονται ασφαλιστικές δικλείδες ε, για την πρόληψη απάτης, κλοπής ταυτότητας ε, και για την αποφυγή καταχρήσεων. Επίσης, η επιγραμμική καταγραφή δεν θα πρέπει να αναρμονίζει τις διατυπώσεις για τη σύσταση εταιρεών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δύο όμως προτάσει οδηγία έπρεπε να μείνουν στο πακέτο και ήταν θετικό αυτό για να έχουμε αποτελεσματικούς κανόνες. για να ε, παρακολουθεί δημιουργία εταιριών γραμματοκιβωτίου για λόγους αφοροαποφυγής, ε, μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και γι' αυτό χαιρόμαστε ε, που είναι το πακέτο αυτό για να μπορούμε έτσι να ξέρουμε συνολικά ποια εργαλεία προβλέπονται. Ε, μάλλον αν δεν ε, ψηφίζουμε υπέρ, απέχουμε, αλλά παρόλα αυτά εκτιμούμε ιδιαίτερα το έργο του κυρίου Σβίφκα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίσω την έναρξη. εγκρινεται Εγκρίνεται 12-1-6. Συγχαρητήρια στον κύριο Ζιρέχκα. Αυτά με τις ψηφοφορίες. Uh, Με την άδειά σας θα προεδρεύσει τώρα ο κύριος Καβαντά ε, για κάποιο διάστημα. Συνάδελφοι, τέλος του διαλύματος, με την άδειά σας να περάσουμε στην, στο σημείο 9, πρόγραμμα δικαιοσύνης. Η συγγήτρια κυρία Χάουταλα, στην οποία θα δώσω το λόγο. Yeah, thank you very much, Chair. Um, as you know, uh, the Parliament uh, uh, about a month ago adopted. Ευχαριστώ πολύ. Όπως ξέρετε, τον προηγούμενο μήνα το Κοινοβούλιο ασχολήθηκε και ενέκρινε το πρόγραμμα των αρχών και αξιών. Τώρα θα ασχοληθούμε με το πρόγραμμα της δικαιοσύνης, το οποίο στόχο έχει να βοηθήσει τους ε, επαγγελματίες του νομικού κλάδου να βελτιώσουν τις δεξιότητες και την ε, αντίληψή τους, την κατανόησή τους του κράτους δικαίου. Είχαμε άρεστες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή και είχαμε έναν πολιτικό τρίλογο, τριμερή διάλογο με την ε, Επίτροπο Γιούροβα που ήταν πολύ θετικός ως προς τα σημεία που ήθελε να προωθήσει το Κοινοβούλιο και στη δική του θέση. Κυρίως θέματα φύλου ε, ως μέρος του νομικού συστήματος και τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και την επίδραση που μπορεί να έχει στη δουλειά των νομικών. Αύριο θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε τις πολιτικές διαπραγματεύσεις και πιστεύω ότι ακόμη μπορούμε να επιδιώξουμε βελτίωση ως προς το πρόγραμμα δικαιοσύνης για να υπάρχει ακόμα περισσότερο περιθώριο για δράση της κοινωνίας των πολιτών. Ιδίω, με την προθυμία που έχει δείξει το Συμβούλιο και η Επιτροπή να πάμε σε αυτό το στόχο, μπορούμε να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα. Είμαι σχετικά ικανοποιημένη και με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου για την ευθυγράμμιση του ρόλου, της διάστασης των φύλων ε, σε όλα τα επίπεδα του νομικού συστήματο μέσω του προγράμματο δικαιοσύνη. Τα πράγματα λοιπόν πάνε καλά και χαίρομαι πολύ γιατί προσωπικώ η Επίτροπο Γιούροβα έχει δείξει μεγάλη αφοσίωση στο σκοπό τη προάσπιση τη ισότητα των φύλων. Καταλαβαίνει ότι η διάσταση του φύλου είναι σημαντική και είναι και πρόθυμη από την αρχή, όπω δήλωσε, να ενισχύσει τη θέση της κοινωνίας των πολιτών στην πρόταση αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι αύριο το απόγευμα θα ξέρουμε περισσότερα. Θα έχουμε τελειώσει και με τον πολιτικό τριμερή διάλογο και εντωμεταξύ βοηθεί και σύμβουλή μας και από την Επιτροπή Γιούρι έχουν εργαστεί σκληρά επί ώρες για να μπορέσουμε να αποπερατώσουμε τα τεχνικά ε, κομμάτια αυτής της πρότασης. Πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Και ελπίζω ότι η πρόταση θα εγκριθεί σύντομα. Ευχαριστούμε κυρία Χάουταλα. Υπάρχουν ε, παρεμβάσεις από τους συναδέλφους. Βλέπω ότι υπήρχε μεγάλη επιτυχία. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε εσεί. Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Κυρία αλλά θέλετε να προσθέσετε τίποτε. Ευχαριστώ. Και τώρα κυρίες και κύριοι σημείο 10, η προστασία των καταγγελόντων. Κυρία Ροζιέρ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από την προηγούμενη ενημέρωση, οι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο συνεχίστηκαν με έναν τρεμερή διάλογο στι 26 Φεβρουαρίου με τεχνικό περιεχόμενο, όπου μπορέσαμε να χτενίσουμε πολλά κομμάτια του κειμένου, μεταξύ των οποίων συμβασμοί για σημαντικά σημεία. Το θετικό είναι ότι υπάρχει διάθεση από την πλευρά των τριών θεσμικών οργάνων να κάνουν ό,τι μπορούν για να ολοκληρωθούν οι διπλωματεύσει πριν τη λήξη τη θητεία. Η διάθεση αυτή λοιπόν υπάρχει, όμως παρά την κινητοποίηση όλων παραμένουν κάποιες δυσκαιρίες. Α σταθούμε πρώτα στι θετικέ πτυχέ. Προχωρήσαμε σε αρκετά σημαντικά σημεία, όπω ε, η σχέση μεταξύ τη οδηγία για την προστασία των καταγγελόντων και τη προστασία των εμπορικών συναλλαγών. Ε, το γεγονό ότι πρέπει κανεί να ε, προστατεύει τους καταγγέλλοντες, να διευρύνει το πεδίο προστασίας τους, λαμβάνοντας όμως υπόψη και τι ε, ενέργειες απαιτούνται για να αποσπαστούν πληροφορίες, θα έχει να κάνει και με την ευθύνη προστασίας των πληροφοριών που καλύπτονται από άλλους κανονισμούς. Η ανάγκη να αποσαφινιστούν οι συνέπειες σε περίπτωση ποινικών ευθυνών, ώστε να παραμείνει και η αρχή της νομιμότητας της διάδοσης πληροφοριών όταν μιλάμε στο για το πεδίο της οδηγίας για την προστασία ενός καταγγέλλοντος. Δηλαδή ε, θα πρέπει να υπάρχει θετική επιρροή, επίδραση, επιπτώσεις από, το, από την πράξη της καταγγελίας αλλά να μην υπάρχουν και άλλε παρενέργειε. Επίση, να μην υπάρξει παραβίαση του επαγγελματικού απορρίτου, που είναι πολύ σημαντικό για την λειτουργία κάποιων επαγγελματικών κλάδων. Ακόμη προχωρήσαμε στο επίπεδο της προστασίας των ε, τρίτων μερών, αυτούς που εμείς ονομάζουμε τους παράγοντες διευκόλυνσης. Δεν έχουμε ολοκληρώσει, έχουμε όμως προχωρήσει. Πρέπει να αποσαφενήσουμε το θέμα της προστασίας της εθνικής ε, προστασίας, της δημόσιας τάξης δηλαδή, για να είμαστε βέβαιοι ότι τα κομμάτια της εθνικής τάξης και ασφάλειας καλύπτονται, χωρίς να διευρυνθεί υπερβολικά η κατηγορία των εξαιρέσεων, των παρεκκλήσεων από αυτή την οδηγία. Επίσης, η διάβλη ε, καταγγελίας. Και αυτό οδηγείται προς αίσιο πέρα, το ίδιο και ως προς τη δημόσια καταγγελία. Τα δύο κείμενα του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σε αυτό το σημείο ε, μάλιστα είναι και πολύ κοντινά. Όμω υπάρχουν κάποιε τεράστιε δυσχέρειε στι δημοτεύσει. Ιδιαίτερα μεγάλε. Εάν τακτοποιηθούν, θα λυθούν ταυτόχρονα. Πρώτη, η ιεράρχηση των διάβλων. Ξέρετε τι συζητήσει έχουν γίνει και στο επίπεδο του Κοινοβουλίου μα. Με διαφορετικέ θέσει να συνεπάρχουν, με μια αυστηρή ιεράρχηση, λιγότερο αυστηρή, με τρει διάβλου καταγγελία, εσωτερικού, εξωτερικού, δημόσιου είναι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις και η θέση του Κοινοβουλίου είναι να μην γίνει ιεράρχηση μεταξύ ε, της ε, εσωτερικής καταγγελίας, δηλαδή στο επίπεδο της επιχείρησης ή εκτός στις αρμόδιες αρχές και να θεωρήσουμε ότι σε μεταγενέστερο στάδιο μπορεί να γίνει και μια δημόσια καταγγελία εφόσον γίνει η πρώτη εσωτερική. Αυτό ήταν η δική μα επιθυμία και η δική μα εντολή. Όμω το Συμβούλιο παραμένει πολύ ε, αμετακίνητο, απαιτώντα μια ε, αυστηρή ιεράρχηση μεταξύ τη εσωτερική και τη εξωτερική καταγγελία. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο περίπλοκα. Και είναι και λίγο περίεργο, γιατί υπάρχει τεράστια συνένεση γύρω από τη θέση του Κοινοβουλίου, μεγάλη υποστήριξη από μη κυβερνητικέ οργανώσει, από του ίδιου του φορεί, από τι συνδικαλιστικέ οργανώσει, το ίδιο το Κοινοβούλιο, και είναι και λίγο παράδοξο, διότι η θέση μα βασίζεται στη σύσταση του Συμβουλίου τη Ευρώπη που έχουν συνυπογράψει όλα τα μέλη του Συμβουλίου τη Ευρώπη, που σήμερα είναι όλα και μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τη Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή. Οπότε δεν γίνεται να υπάρχουν τόσο αποκλίνουσε θέσει ε, για θέματα στα οποία έχουν ήδη προσυμφωνηθεί. Αυτά ω προ τι διαπραγματεύσει. Άλλη δυσχέρεια, το θέμα του τι γίνεται με μικρότερε σημασίε καταγγελία, ίσονο σημασία, αυτό μπορεί να επιληθεί αν λύσουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα και εκεί που υπάρχει και μεγάλη διαφωνία είναι το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Ε, μια προσέγγιση όπου φέρνει ε, αντιδιαμετρικά αντίθετους στις προσεγγίσεις του στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το θέμα του εργατικού δικαίου δηλαδή και τη εταιρική προστασία. Το Συμβούλιο θέλει να περιοριστεί εδώ το πεδίο. Και το ίδιο και για το παράρτημα που ορίζει μια σειρά από ευρωπαϊκά κείμενα από από τη οδηγία και ε, αναφέρονται ενδεικτικά. Το, κοινοβούλιο, το Συμβούλιο όμω θεωρεί ότι αυτό είναι περιοριστικό και μας δεσμεύει. Εκεί λοιπόν υπάρχει ακόμα πολλή συζήτηση. Διάθεση να προχωρήσουμε υπάρχει. Υπάρχουν ε, βαθιές διαφωνίες βεβαίως, δύσκολο να επιληθούν και να εξομαλυνθούν, αλλά θέλουμε να προχωρήσουμε, το ξανάπα. Ας παραμείνουμε συγκρατημένοι αισιόδοξοι για την ε, δυνατότητά μας να πετύχουμε ολοκλήρωση της εξέτασης του θέματο. Ε, έχουμε μέχρι τα μέσα Μαρτίου 10 μέρες περίπου για να τα καταφέρουμε. Θα ε, επιταχύνουμε Ευχαριστώ όλους τους, όλα τα μέλη της δημοτευτικής ε, ομάδας και τους σκιώδεις εισηγητές και τους συνεργάτες μας για τα τεχνικά θέματα. Ελπίζω ότι θα πετύχουμε συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Ποιος έχει ζητήσει το λόγο, κανένας. Εκπλήσωμε. Ή τέλο πάντων, μάλλον τίποτα δεν με εκπλήσει πια σε αυτή τη φάση. Με την άδειά σα, ε, κύριε Συγγήτρια, αγαπητή συνάδελφοι, να πω εγώ κάτι ω κοιόδη συγγητή. Ε, μπορώ να κάτσω και στην πλανή καρέκλα, αν θέλετε. Τέλο πάντων, καταρχά θέλω να στηρίξω τη δήλωση τη συγγήτρια ε, σε ό,τι αφορά τη θέση του Κοινοβουλίου, που είναι πραγματικά ισορροπημένη, χωρίς όμως να στερεί το κείμενο από το νόημά του και νομίζω ότι το είπατε πολύ. Ε, συχνά στην ομιλία σε τρία θεσμικά όργανα ότι αυτή είναι η οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε. Μια παρατήρηση είναι ότι σε ό,τι αφορά εμένα τουλάχιστον εμείς είμαστε προσιλωμένοι στη θέση του Κοινοβουλίου αλλά κυρίως σε δύο θέματα που εγώ θέλω να αναφέρω. Το πρώτο είναι η διατήρηση του παραρτήματος με ενδεικτική αξία και το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, προαιρετικός χαρακτήρας αυτών των διάβλων καταγγελίας. τι βλέπω ότι υπάρχει μια ισχυρογνωμοσύνη. Θα δούμε τι θα γίνει στις 7 ε, τα απόγευμα σήμερα. Μέχρι στιγμή βλέπουμε ισχυρογνωμοσύνη από πλευράς του Συμβουλίου και αυτό δεν ε, κάνει σε κανέναν χάρη ούτε στι υπηρεσίε ούτε στου καταγγέλλοντε. Αυτού δηλαδή οι οποίοι καταγγέλουν και πολλέ φορέ βάζουν σε κίνδυνο την φήμη, την υπόλοιψη και την ε, σταδιοδρομία του για να καταγγείλουν κάτι το οποίο θεωρούν ότι είναι άκρο επιζήμιο για το δημόσιο γενικό συμφέρον. Δεν το κάνουν για το μισθό του, για την πραγωγή του. Δεύτερον, σε αυτές τις συνθήκες, αυτές τις μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υποκαθιστούν τη δράση των εθνικών αρχών, των δημόσιων αρχών, που θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα, δεν είναι σε επιχειρήσει βέβαια. Άρα μόνο οι πάλι των επιχειρήσεων, τέλο πάντων αυτοί που έχουν κάποια σχέση με αυτού, μπορούν να παρέμβουν. Και επομένω, από αυτέ τι συνθήκε, δεν θα πρέπει να αρκεστούμε στον εσωτερικό διάβλο, ούτε και να γίνει αυτό υποχρεωτικό. Πρέπει να είναι προαιρετικό. Πρώτη επιλογή, το α μικρό, εσωτερικό διάβλο τη επιχείρηση και β μικρό, που είναι και πιο ε, πιθανό, εξωτερική αρχή, εξωτερική της επιχείρησης αρχή, η οποία θα ερευνά το βάσιμο ή το κατά πόσο υπάρχει κακοπιστία ή ε, δυσφήμιση εκ μέρους του καταγγέλλοντος. Αυτή δεν είναι η άποψη του Συμβουλίου αυτή τη στιγμή, ε, διότι αν είναι κάτι σοβαρό, τις περισσότερες φορές ε, το ξέρει η, η αρχή και αν δεν ε, κάνει κάτι για να πάψει αυτή τη λειτουργία, σημαίνει ότι δεν θέλει να πάψει αυτό. Σας υπενθυμίζω τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στο Κοινοβούλιο με τα λογισμικά που επηρέαζαν τις τιμές ε, των εκπομπών καυσαερίων, τα οχήματα. Άρα, να βλέπουμε αν είναι ε, καλή πίστη και αν είναι κάτι παραδεκτό και μετά βλέπουμε τον εσωτερικό διάβλο ή τον εξωτερικό. Και αν δεν λειτουργεί τίποτα, από τα δύο έχουμε τους ε, δημοσιογράφους, τον τύπο. Το κοινοβούλιο δεν ξέρω γιατί έχει πεισμώσει. Δύσκολα, δυσεξήγητα τα κίνητρα. Δεν ξέρω αν είναι φόβος και ελπίζω να μην είναι κακή πίστη. Ε, μακάρι να μπορούσαν να μετακινηθούν. Αυτά είχα να πω. Και συγγνώμη που καταχράστηκα τι θέσει του Πρόεδρου για να εκφράσω άποψη ενό εισηγητού. Νομίζω πάντω ότι η πραγματευτική μα ομάδα είναι ενωμένη ε, για ένα θέμα πολύ σημαντικό που είναι βέβαια και δύσκολο. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν το λόγο, όχι. Η Κομισιόν, κυρία Ροζιέρ, θέλει να προσθέσει κάτι. Η κυρία Κάφμαν ήθελε το λόγο. πάρα πολύ σύντομη θα είμαι. Άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά και βεβαίω άκουσα πολύ προσεκτικά και την εισηγήτριά μας ε, και όλα αυτά που περιέγραψε, κυρίως όσον αφορά το θέμα των ε, διαφόρων καναλιών Νομίζω λοιπόν ότι ως κοινοβούλιο ε, πρέπει να λάβουμε θέση. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό το θέμα. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ενθαρρύνω την εισηγήτρια να μην ενδώσει γιατί μερικές φορές ε, ε, δεχόμεθα πιέσει, ε, πολιτική πίεση, πίεση χρόνου, αλλά το θέμα είναι να μην καταλήγουμε ε, στο να πληρώνουμε ένα πολύ ψηλό τίμημα για να μπορούμε να επιτύχουμε ενότητα. να μπορούμε να πούμε και ότι όχι δεν συμφωνούμε μετά από όλα αυτά που άκουσα, προς τα εκεί κατευθύνεται η όλη υπόθεση. Από την άλλη βέβαια ε, είμαι πρόθυμη να μοιραστώ την αισιοδοξία της εισηγήτριας αλλά ο συμβασμός χάρη και μόνον του συμβασμού αυτό ε, νομίζω ότι ε, είναι μια πολύ απλουστευτική αντιμετώπιση και δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα των whistleblowers που εκπροσωπούμε. Δεν θέλει κανείς άλλος να λάβει το λόγο. Και πάλι ο Σκιώδης, και σε το συγγνώμη, επειδή μου δώσετε μια ιδέα, κυρία Κάφμαν. Δεν είναι καλός υπολογισμό ε, να θέλουμε να ιεραρχήσουμε τα πράγματα όπως το κάνει το Συμβούλιο. Καλά, σίγουρα υπάρχει ε, μια σύνθεση των, με, του Συμβούλου. Και χειρότερη αυτή τη Ένωση τελικά είναι τα μέλη. Αλλά τέλο πάντων, το ξέρουμε αυτό. Μην δημιουργούμε όμω πάθη και παρακολύουμε την καταγγελία. Οι καταγγέλλοντες δεν καταγγέλουν έτσι ε, για ψηλουπίδημα και αν το κάνουν ε, θα την πατήσουν μετά. Αλλά αν το κάνουν συνήθως είναι για κάτι σοβαρό. Και νομίζω ότι σε αυτήν την περίπτωση είναι φυσικά να πούμε ότι θα έχουμε ή την εσωτερική καταγγελία ή την εξωτερική αρχή. Γιατί αλλιώς ο καταγγέλων θα πάει στον τύπο και θα έχουμε τα σκάνδαλα και τον υποδάβληση των παθών και τα λοιπά. Θα το σκεφτούμε. Συγγνώμη που ξαναπήρα το λόγο να συμπληρώσω. Ε, κύριε Ροζιέ, θέλει το λόγο. Ναι. Να συμπληρώσω κάτι. Έτσι για να βάλουμε λίγο τον κοινό νου ξανά στη συζήτηση. Το επιχείρημα για αυτή την αυστηρή ιεράρχηση νομίζω είναι ο παράλογος φόβος. ότι θα γεμίσουμε από καταγγέλλοντες και θα ε, κατακλείζονται οι δημόσιες ε, αρχές από τέτοιου είδους καταγγελίες. Γι' αυτό και είναι καλό και ενάρετο να θέλουν οι επιχειρήσεις να οργανώσουν εσωτερικούς διάβλους ε, ε, για τις καταγγελίες αυτές. Όμως συχνά δεν υπάρχει αυτή η υποχρέωση, δηλαδή εσωτερικός ή εξωτερικός διάβλος και το λέει και η μελέτη αντικτύπου της Κομισιόν ότι όταν οι διάβλοι καταγγελίας είναι, ε, υπάρχουν μέσα στην επιχείρηση και ο καταγγέλων ε, καλείται να αποφασίσει ποιος είναι ο καλύτερος διάβλος στις 90% των περιπτώσεων ε, πάνε στο εσωτερικό διάβλο αρκεί να είναι αποτελεσματική και να λύνεται έτσι το πρόβλημα. 90% δηλαδή πηγαίνουν στους εσωτερικούς διάβλους. Όταν είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό, χρησιμοποιείται αυτή η άμεση καταγγελία ε, στο 10% των περιπτώσεων. Είναι κρίμα λοιπόν να βάλουμε την ρητή υποχρέωση και ουσιαστικά να μην τους ε, παραχωρούμε την προστασία που πρέπει να τους εξασφαλίζουμε. Γιατί μπορεί να υπάρξουν ε, αντίπεινα. Αλλά το θέμα είναι ότι αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα δεν θα είναι αποτελεσματική η καταγγελία. Δεν θέλει κανείς το λόγο την Κομισιόν. Ωραία. Έχουμε λοιπόν εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες και θα συνεχίσουμε και κλεισμένο των θυρών. Όσοι δεν έχουν λόγο να βρίσκονται εδώ, παρακαλώ να αποχωρήσουν.